και κύριοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Πριν από 26 χρόνια, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο δεύτερος εκφώνησε ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η ομιλία του αποτέλεσε ορόσημο στο δρόμο για την πτώση του σιδηρού ε, παραπετάσματος και για τη διάνοιξη της ε, οδού για την επανένωση στην Ευρώπη. Σήμερα απευθύνεστε εσείς, Πάπα Φραγκίστου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μέλη που εκπροσωπούν πάνω από 500 εκατομμύρια πολιτών και 28 χώρες μέλη. Οι βουλευτές του Κοινοβουλίου αντανακλούν την ποικιλομορφία της Ευρώπης. Την τελευταία εξαετία η Ευρώπη έζησε μια δραματική κρίση ανευπροηγουμένου με βαριές συνέπειες. Ιδιαίτερα τραγική είναι η απώλεια εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στα θεσμικά τους όργανα και στους θεσμούς τους, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Και αυτή η απώλεια εμπιστοσύνη είναι τεράστια. Χωρίς εμπιστοσύνη όμως δεν μπορεί καμία ιδέα, για να μην πω κανένας θεσμός, να ε, υφίσταται στο δίνεκε. Γι' αυτό απαιτείται συνεργασία όλων των δυνάμεων έτσι ώστε να ανακτηθεί η χαμένη αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Προς την κατεύθυνση αυτή εργάζονται τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η Καθολική Εκκλησία σε μεγάλο βαθμό χέρι-χέρι. Οι αρχές της ε, ανεκτικότητας, του σεβασμού, της ισότητας, ε, της ε, ειρήνης και της αλληλεγγύης είναι αξίες και τμήματα της κοινή μας εντολής η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρεσβεύει το ε, να συνεπάρχει κανείς και όχι να είναι ένας απέναντι στον άλλον, τη συμπερίληψη και όχι τον αποκλεισμό, την ένταξη. Οι νέοι θα πρέπει να βρουν εργασία και θέσεις στην κοινωνία, οι μετανάστες αναζητούν για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους ένα καλύτερο μέλλον. Ο κόσμος φεύγει από πολέμους και καταστροφές και ολέθρους και ζητά σε εμάς άσυλο και προστασία είτε πρόκειται για την κοινωνική δικαιοσύνη ή για την άνηση κατανομή ε, των ευκαιριών και του πλούτου, είτε πρόκειται για την κατάσταση των πιο ηλικιωμένων στην κοινωνία μας, είτε πρόκειται για πολέμους και σειράξεις στην άμεση γειτονία μας, αλλά και πέρα από αυτά, είμαστε ενώπιον κοινών προκλήσεων όλοι. Αγιότατε, τα λόγια σας έχουν τεράστια σημασία. Όχι μόνο διότι είστε ε, ο θρησκευτικό ηγέτης ε, ε, για τους καθολικούς που είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο στον κόσμο. Αλλά έχουν μεγάλη σημασία τα λόγια σας γιατί μας αφορούν όλους και απευθύνονται σε όλους μας. Και έχουν ισχύ για όλους μας, διότι τα θέματα που διαπραγματεύεστε μας αφορούν όλους και μας συγκινούν όλους. Είναι παγκόσμια, οικουμενικά αυτά τα θέματα. Τα λόγια σας δίνουν προσανατολισμό σε καιρούς που έχουμε χάσει την πηξίδα μας. Το μήνυμά σας για την ειρήνη και το διάλογο, ε, για την ακαιρεότητα και την ευθύνη του ενός για τον άλλον, για την αλληλεγγύη και για τη συμβίωση, μας καθιστούν σαφές ότι έχουμε κοινούς ε, στόχους, κοινέ προκλήσεις και θα πρέπει από κοινού να τις αντιμετωπίσουμε. Ότι ενωμένοι είμαστε πιο ισχυροί από ότι ο καθένας μόνος του. Το δικό σας μήνυμα είναι πάρα πολύ ευρωπαϊκό, διότι ακριβώς ε, σε αυτό το μήνυμα βασίζεται η ίδια ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Και η δική σας ιστορία, Γιώτατε, είναι ευρωπαϊκή. Είναι ιστορία μιας οικογένειας που εγκατέλειψε την Ευρώπη για να ζήτησε μια νέα πατρίδα, την οποία και βρήκε στην Νότια Αμερική. Είναι ιστορία ενός Πάπα, ε, ο οποίος προέρχεται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού και γυρνάει από τα πέρατα του κόσμου στην Ευρώπη για να μεταρρυθμίσει την εκκλησία του και να ηγηθεί των πιστών. Είναι μια ιστορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να βοηθήσει την Ευρώπη να αποτελέσει παράδειγμα και υπόδειγμα για να μεταρρυθμιστεί η Ευρώπη και να ανανεωθεί. Σας ευχαριστώ εξ όλων των συναδέλφων μου που αποδεχθήκατε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρευρίσκεστε σήμερα ενώπιον μας. Αποτελεί τιμή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και προνόμιο η ευκαιρία που έχει να μπορεί να σας ακούσει. Αγιότατε Πάπα Φραγκίσκο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Αντιπρόεδροι, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, όλοι όσοι εργάζονται σε αυτό το ημικύκλιο, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να πάρω το λόγο ενώπιον αυτού του θεμελιώδους θεσμού για τη ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ μέσω ημών στους πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες που εκπροσωπούν τις 28 χώρες μέλη. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη θα ήθελα να εκφράσω προς εσάς κύριε Πρόεδρο του Κοινοβουλίου για τα θερμά λόγια καλωσορίσματος τα οποία μου απευθύνατε εξ ονόματος όλων ε, όσοι βρίσκονται στην ε, Ολομέλεια. Η επίσκεψή μου αυτή έρχεται 25 και πλέον χρόνια μετά από αυτήν του Ιωάννη Παύλου Δευτέρου. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν πλέον τα αντιτιθέμενα μπλοκ τα οποία τότε χώριζαν τον, ε, την Ήπειρο στα δύο. Και σιγά σιγά ε, καλύπτεται η επιθυμία η Ευρώπη μέσα από ελεύθερες και κυρίαρχες ε, οργανώσεις και θεσμούς να μπορέσει να φτάσει σε αυτές ε, τις ε, διαστάσεις που τις είχε δώσει η γεωγραφική δόμηση αλλά ακόμα περισσότερο η ίδια η ιστορία δίπλα σε μια ευρεία ή ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει βέβαια και ένας κόσμος πιο περίπλοκος ο οποίος βρίσκεται διαρκώς εν κινήσει. Ένας κόσμος ο οποίος είναι όλο και περισσότερο διασυνδεδεμένος και παγκοσμιοποιημένος και επομένως όλο και περισσότερο ευρωκεντρικός. Σε μια πιο εκτεταμένη ένωση και που θα έχει μεγαλύτερη επιρροή ε, πάντα θα πρέπει να βάζουμε και μια ε, εικόνα μιας Ευρώπης λίγο γερασμένης η οποία αισθάνεται λιγότερο πρωταγωνίστρια ε, σε ένα περιβάλλον που συχνά ε, την βλέπει με καχυποψία και με έλλειψη εμπιστοσύνης πολύ συχνά. Απευθύνομαι σε εσά σήμερα ως ποιμήν και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να απευθύνω σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα μήνυμα ελπίδας και ενθάρρυνσης. Ένα μήνυμα ελπίδας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην πεποίθηση ότι μπορούν οι δυσκολίες να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ενότητα και θα μπορέσουν να νικήσουν τους φόβους της Ευρώπης μαζί με ολόκληρο τον κόσμο και επίσης ε, ε, ελπίδα στον ε, Κύριο ο οποίος μετατρέπει το καλό σε κακό και το θάνατο σε ζωή. Ενθάρρυνση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τις πεπιθήσεις των πατέρων που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι ήθελαν ένα μέλλον που θα βασίζεται σε υπέρβαση των διαφορών και κοινωνία μεταξύ όλων των πολιτών και της Ευρώπης. Στο κέντρο αυτού του Εβραίου πολιτικού και φιλόδοξου πολιτικού προγράμματος βεβαίως υπήρχε η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Όχι τον άνθρωπο ως πολίτη, αλλά ε, ε, ούτε και ως ε, πολιτικού υποκειμένου, αλλά σαν ένα άτομο το οποίο διαθέτει υπερβατική αξιοπρέπεια. Θέλω πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω αυτήν την μεγάλη ενότητα που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο λέξεις, υπέρβαση και αξιοπρέπεια. Η αξιοπρέπεια είναι μια λέξη κλειδί η οποία χαρακτηρίζει το, ε, την περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ε, η ιστορία μας βεβαίως διακρίνεται από την ε, ανθρωποκεντρικότητα και καταφέρεται εναντίον κάθε μορφής βίας και διακριτικής μεταχείρισης η ε, αντίληψη της ε, ε, ικανότητας αυτής των ανθρώπων έχει περάσει μέσα από ένα μακρύ δρόμο, μέσα από θυσίες και μέσα από δυσκολίες οι οποίες δημιούργησαν αυτήν την έννοια της άρρηκτης πραγματικότητας που διαμόρφωσε αυτήν την ιδέα ότι όχι μονάχα μέσα από την ιστορία αλλά και κυρίως στην ευρωπαϊκή σκέψη ε, η οποία βασίζεται ακριβώς στην πλούσια συνάντηση ε, πολλών στοιχείων που προέρχονται από την Ελλάδα, από τη Ρώμη, από στοιχεία γερμανικά, κελτικά, σλαβικά και από τον χριστιανισμό που διαμόρφωσε σε βάθος αυτήν την έννοια του ατόμου. Σήμερα η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, παίζει κεντρικό ρόλο στην δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε ε, να ε, αξιοποιηθεί περισσότερο και να προωθηθεί η αξιοπρέπεια του ατόμου και στις σχέσεις μεταξύ άλλων ανθρώπων και στις σχέσεις με άλλες χώρες. Πρόκειται βεβαίως για μια αξιοθαύμαστη δραστηριότητα. Παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα πολλές περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σαν σαν ε, αντικείμενα των οποίων το λειτουργικό ή το λογισμικό μπορεί να προγραμματιστεί και τα οποία τα πετάμε όταν δεν ε, χρησιμεύουν πλέον γιατί είναι μεγάλοι, γιατί είναι ε, άρρωστοι ή ηλικιωμένοι. Πραγματικά ποια αξιοπρέπεια μπορεί να υπάρχει όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα να εκφράσει κανείς είτε τη σκέψη του είτε την πολιτική του πίστη. Ποια αξιοπρέπεια μπορεί να υπάρχει χωρίς καθαρό νομικό πλαίσιο το οποίο θα περιορίσει την κυριαρχία της δύναμης ε, και ε, της εξουσίας. Ποια αξιοπρέπεια μπορεί να έχει ένας άνδρας ή μια γυναίκα που υφίσταται κάθε είδους διακριτική μεταχείριση, ποια αξιοπρέπεια μπορεί να βρει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει φαγητό ή δεν έχει τα ελάχιστα έτσι ώστε να επιβιώσει ή που χειρότερο ακόμα δεν έχει αυτήν την εργασία η οποία μπορεί να του δώσει αξιοπρέπεια. η πρόθεση αξιοπρέπεια του προσώπου σημαίνει ε, ότι καταλαβαίνουμε ότι αυτό το πρόσωπο έχει αναπαλωτρίωτα δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί να του στερήσει κανείς ε, με δική του απόφαση και κυρίως όχι λόγω οικονομικών συμφερόντων. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην πέσουμε σε παρεξηγήσεις οι οποίες μπορούν ε, να ξεκινήσουν από μια ε, άσχημη ε, κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πράγματι τίνουμε να έχουμε διαρκώς περισσότερες διεκδικήσεις όσον αφορά τα ατομικά δικαιώματα, τα εξατομικευμένα δικαιώματα και ατομιστικά δικαιώματα, δηλαδή ενός ατόμου που τα δικαιώματά του είναι σχεδόν, αντιμετωπίζονται σχεδόν ως μία μονάδα ε, η οποία δεν δείχνει καμία ευαισθησία προς τις άλλες μονάδες που αποτελούν την κοινωνία. Στην ε, ε, ιδέα του δικαιώματος φαίνεται ότι ξεχνούμε να βάλουμε την απαραίτητη έννοια δίπλα του καθήκοντος. Δεν λαμβάνουμε υπόψη επομένως ότι κάθε ανθρώπινο «ον» είναι συνδεδεμένο με το κοινωνικό κοινωνικό του πλαίσιο και ότι οι υποχρεώσεις του ε, και τα καθήκοντά του συνδέονται με τα άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις των υπολείπων μελών της ιδίας κοινωνίας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ζωτική σημασία ε, να ε, προσπαθήσουμε σήμερα να βρούμε και να εμβαθύνουμε σε μία κουλτούρα, σε ένα πολιτισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων που με σοφό τρόπο με, να λαμβάνει υπόψη του την ατομική διάσταση ή μάλλον να πω καλύτερα την προσωπική διάσταση σε σχέση όμως με την κοινωνία ε, όλων ημών που αποτελούμε την υπόλοιπη κοινωνία. Πραγματικά σήμερα δεν υπάρχει αρμονική διασύνδεση ανάμεσα στο εγώ και στο εμείς ε, και αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή βιαιοτήτων και σειράξεων. Το να μιλήσει κανείς για την υπερβατική αξιοπρέπεια του ανθρώπου σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνει έκκληση στην φύση του, στην εγγενή του δυνατότητα και ικανότητα να διαχωρίζει το καλό και το κακό. Ε, από αυτήν την πηξίδα την οποία έχει χαράξει ο Θεός στις ε, καρδιές μας. Να ε, κοιτάμε δηλαδή τον κόσμο, όχι μονάχα ε, τον άνθρωπο και το άτομο, το, το πρόσωπο, όχι μονάχα σαν ένα απόλυτο, αλλά και σαν με ένα μέλος μιας κοινωνικής κοινωνίας. Γιατί διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε αυτήν την τρομερή μοναξιά. Ακριβώς αυτή τη μοναξιά στην οποία οδηγείται το άτομο όταν ε, δεν έχει άλλους δεσμούς. Αυτό ισχύει περισσότερο για τους ηλικιωμένους ας πούμε, τους οποίους εγκαταλείπουμε ή ισχύει και για τους νέους οι οποίοι αισθάνονται ότι ε, δεν έχουν πλέον κανένα μέλλον. Το βλέπουμε, το βλέπουμε στους ε, πολλούς φτωχούς που ζουν πλέον στις χώρες μας. Το, το βλέπουμε και στο χαμένο βλέμμα των μεταναστών που έρχονται στις χώρες μας προσπαθώντας να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η μοναξιά έχει οξυνθεί βεβαίως από την οικονομική κρίση τα αποτελέσματα της ε, οποίας ακόμα παράγουν ε, πολύ αρνητικά αποτελέσματα από κοινωνικής απόψεως. Μπορούμε επίσης να διαπιστώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια μαζί με την διαδικασία διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, αυξήθηκε και η καχυποψία από πλευράς των πολιτών προς θεσμούς, η δυσπιστία συγγνώμη, ε, προς θεσμούς οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να αγγίξουν τις ευαισθησίες των κρατών μελών και των πολιτών και που πολλές φορές θεωρούν ότι παίρνουν αποφάσεις ακόμα και επιζήμιες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μια γενική αίσθηση κόπωσης, γύρανσης μιας Ευρώπης η οποία δεν έχει πλέον ζωτικότητα και δεν μπορεί ε, να είναι γόνιμη. Τα μεγάλα ιδεώδη τα οποία έμπνευσαν την ε, Ευρώπη φαίνεται ότι έχουν χάσει την ε, ισχύ τους προς όφελος κάποιων πιο γραφειοκρατικών αντιμετωπίσεων. Εδώ θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε και τρόπους ζωής εγωιστικούς ε, που βασίζονται στη χλειδί, μία χλειδί η οποία συχνά ε, και δεν μπορεί να συντηρηθεί αλλά και συχνά δείχνει αδιαφορία, αδιαφορία απέναντι στο γύρο κόσμο κυρίως όσον αφορά τους πιο φτωχούς διαπιστώνουμε με θλίψη ότι υπερέχουν τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα τα οποία βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της ε, ε, πολιτικής συζήτησης προς ζημία ε, μιας αυθεντικής ανθρωπολογικής διάστασης. Το ανθρώπινο «ον» όλο και περισσότερο γίνεται ένα απλό γρανάζι σε ένα μηχανισμό ο οποίος βασίζεται μονάχα στον καταναλωτισμό. Και όταν η ζωή δεν μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το μηχανισμό και δεν είναι πλέον ένα χρήσιμο γρανάζι, τότε πετάμε τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι, τους ανθρώπους ε, που δεν χρειάζεται πλέον να τους ε, κρατήσουμε σε ζωή γιατί δεν μπορούν πλέον ε, να θεραπευθούν ή ακόμα και τα παιδιά. Αυτή είναι η μεγάλη παρανόηση η οποία ε, προκύπτει ε, όταν ε, υπερισχύει η απολυτότητα της τεχνικής και δημιουργείται μια σύγχυση ανάμεσα στο μέσο και το σκοπό. Και βεβαίως έτσι φτάνουμε στην κουλτούρα του αναλώσιμου και του απελπισμένου καταναλωτισμού. Αντιθέτως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία ε, της ανθρώπινης ζωής, ε, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που βεβαίως δεν μπορεί να αποτελέσει είτε αντικείμενο ε, εμπορίας είτε ανταλλαγής. Εσείς ως κοινοβουλευτικοί καλείστε να επιτελέσετε σημαντικό έργο, έστω και αν μερικές φορές μπορεί να φαρεί ανώφελο. Εσείς θα πρέπει να λάβετε υπόψη, να αναλάβετε την τροτότητα, την ευαλωτότητα των λαών και των ανθρώπων. Θα πρέπει ε, να βοηθήσετε με ε, δύναμη αλλά και με τρυφερότητα αυτούς τους ανθρώπους. Να φροντίσετε έτσι ώστε από ένα μοντέλο το οποίο οδηγεί σε αυτήν την ε, κουλτούρα του αναλώσιμου ε, να ε, αναλάβετε με τρυφερότητα τους ανθρώπους. Και αυτό ακριβώς σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις προσδοκίες, τις ελπίδες των ανθρώπων. Να λάβετε υπόψη σας αυτούς τους πιο περιθωριακούς που περισσότερο χρειάζονται την αξιοπρέπεια. Πώς μπορούμε να ξαναδώσουμε ελπίδα στο μέλλον, έτσι ώστε ξεκινώντας από τις νέες γενναίες να ξαναβρεθεί αυτή η εμπιστοσύνη έτσι ώστε ε, να ε, ακολουθηθούν τα μεγάλα ιδεώδη της ε, ενωμένης και ειρηνικής Ευρώπης, της δημιουργικής Ευρώπης, η οποία επιχειρεί, η οποία όμως σέβεται και τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβάνοντας υπόψη και γνωρίζοντας τις δικές της υποχρεώσεις. Για να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, επιτρέψτε μου να σας δώσω μία εικόνα. Ένα από τα, μία από τις φημισμένες τοιχογραφίες του του Ραφαήλ που βρίσκονται στο Βατικανό ε, αντιπροσωπεύει τη λεγόμενη Σχολή των Αθηνών. Στο κέντρο του υπάρχει ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. Ο πρώτος δείχνει με το δάχτυλο προς τα ψηλά, προς τον κόσμο των ιδεών, μπορούμε να πούμε ότι δείχνει προς τον ουρανό. Ο δεύτερος ε, ε, δείχνει μπροστά με το δάχτυλό του προς την πραγματικότητα, τη συγκεκριμένη αυτή πραγματικότητα προς τη γη. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα η οποία καλά περιγράφει την ε, Ευρώπη και την ιστορία της, ε, η οποία έχει δημιουργηθεί από την διαρκή συνάντηση μεταξύ της γης ε, και του ουρανού, όπου ο ουρανός πάντα έδειχνε την υπέρβαση και το άνοιγμα προς το Θεό και όπου η γη πάντα εκπροσωπούσε τις πρακτικές ικανότητες και την συγκεκριμένη δυνατότητα αντιμετώπισης καταστάσεων και προβλημάτων. Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την ε, επανέβραση αυτού του ζωτικού και αδιάρρηκτου δεσμού που υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα αυτά τα δύο στοιχεία. Μία Ευρώπη η οποία θα είναι ικανότερη να ανοιχτεί προς αυτήν την υπερβατική διάσταση τη ζωή. Μία Ευρώπη η οποία χάνει δυστυχώ σιγά σιγά αυτό το ουμανιστικό ανθρωπιστικό ε, πνεύμα στο οποίο όμως θα πρέπει να βασιστεί. Ακριβώς εδώ θα ήθελα εγώ ε, να πω ότι πρέπει να ε, υπάρξει ένα νέο άνοιγμα προς αυτήν ε, την διάσταση, την υπερβατική του ανθρώπου και πιστεύω ότι αυτό δεν αναφέρεται μονάχα στον χριστιανισμό και την το κληροδότημα το οποίο έχει αφήσει προς ε, την ε, ε, Ευρώπη αλλά πιστεύω ότι αυτή είναι η συμβολή η οποία θα αποτελέσει βασική συμβολή για το μέλλον και αυτή η συμβολή, η συμβολή συγγνώμη, δεν αποτελεί κανένα κίνδυνο για την λαϊκότητα, κοσμικότητα των κρατών. Αντιθέτως βασίζεται σε αυτές τις αρχές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε αρχές όπως είναι η αλληλεγγύη, αμοιβαία αλληλεγγύη ε, όπως είναι η επικουρικότητα, ε, δηλαδή μία ε, αλληλεγγύη και μία κεντρική ανθρωπιστική αντιμετώπιση η οποία μπορεί να αποτελέσει ακριβώς το κέντρο αυτών των αποφάσεων. Ακριβώς εδώ θα ήθελα να σας πω ότι για μία ακόμα φορά ε, σας λέγω ότι η Άγια Έδρα είναι διαθέσιμη ε, για έναν ανοιχτό και καρποφόρο διάλογο ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη γενικά θα πρέπει να αποθυσαυρίσει όλες αυτές τις δυνατότητες τις οποίες δίνουν όλες οι γνώσεις και οι ρίζες ακόμα και της Εκκλησίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό, το κενό των ιδεών το οποίο ε, στη λεγόμενη Δύση ε, διαπιστώνουμε σήμερα και που μονάχα ε, ο Θεός μπορεί να καλύψει γιατί η εξήμνηση και όχι η λύθη του Θεού οδηγεί συγγνώμη, η λύθη του Θεού και όχι η εξήμνησή του οδηγεί στι ακρότητες και, και τη βία. Δεν είναι δυνατόν να λησμονήσουμε τις πολλέ αδικίες και τους διωγμούς που πλήττουν καθημερινά τις ε, ε, μειονότητες, θρησκευτικέ μειονότητες, κυρίως δε τους χριστιανούς σε διάφορα μέρη του κόσμου. Κοινότητες και άνθρωποι που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν βαρβαρότητες και ε, βία, που εκτοπίζονται από τις χώρες τους, από τα σπίτια τους, που αποκεφαλίζονται, που καίγονται ενώ οι περισσότεροι σιωπούν σε μια συνένοχη σιωπή. Το σλόγγαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ενότητα στη διαφορετικότητα. Αλλά ενότητα δεν σημαίνει πολιτική ομοιογένεια ή οικονομική ή πολιτιστική ε, ή ομοιογένεια σκέψης. Στην πραγματικότητα κάθε αυθεντική ενότητα ε, ζει από, την, ε, από τον πλούτο των διαφοροτήτων που την συστήνουν ακριβώς αυτή η πολυφορμία, η ε, πολυμορφία μπορεί να οδηγήσει ε, σε αυτόν τον εμπλουτισμό. Κατά αυτή την έννοια θεωρώ ότι η Ευρώπη είναι μία ε, οικογένεια λαών που μπορούν να αισθανθούν και πρέπει να αισθανθούν κοντά ε, στους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς εάν αυτοί καταφέρουν να συνδέσουν ακριβώς αυτήν την ειδική πραγματικότητα του καθενός με την ενωτική πολυμορφία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις κοινέ ρίζες στην ιστορία απελευθερωνόμενοι από όλες ε, τις φοβίες ε, ή τις προσπάθειες εγχειρηματοποίησης και βεβαίως ε, σημαίνει το να βάλουμε τον άνθρωπο στο κέντρο ε, της δραστηριότητάς μας σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα δικαιώματα και των ατόμων και των λαών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη βέβαια και τις ιδιαιτερότητες του καθενός γιατί αυτές αποτελούν μεγάλο ε, πλούτο θα πρέπει να θυμίσουμε ε, την, την ίδια την αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται στις αρχές ε, της επικουρικότητας ε, και της αλληλεγγύης έτσι ώστε να υπερισχύσει η ουσιαστική βοήθεια και έτσι ώστε εμψυχωμένοι να μπορέσουμε να οδηγηθούμε προς την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Σε αυτήν την δυναμική της ε, ε, ε, ιδιαιτερότητας και της ενότητας. Κύριοι και κυρίες Ευρωβουλευτέ, θα πρέπει να λάβετε υπόψη και την απέτηση να παραμείνει ζωντανή η δημοκρατία στην Ευρώπη, η δημοκρατία των λαών στην Ευρώπη είναι σαφές ότι ε, η ε, πραγματική απόφαση, ότι κάποιες αποφάσεις ε, που αφορούν παγκοσμιοποιημένες αποφάσεις μπορούν να αποδυναμώσουν ένα δημοκρατικό σύστημα. Διατρέχουμε λοιπόν τον κίνδυνο να ζήσουμε στην, ε, ε, στο, στο πνεύμα του λόγου μονάχα και της σοφιστίας και τελικά να μπερδέψουμε την πραγματικότητα της ε, δημοκρατίας με ένα νέο πολιτικό νομιναλισμό. Θα πρέπει να διατηρήσουμε πραγματικά ε, την ε, ε, ιδέα της δημοκρατίας μακριά από αγγελικούς πουρισμούς, από απολυταρχίες του σχετικού, από ανιστόρητους φονταμενταλισμούς, από ηθικολογίες χωρίς καλοσύνη και από διαλογισμούς χωρίς σοφία. Θα πρέπει να αποφύγουμε το γεγονός ότι η πραγματική τους ε, δυνατότητα έκφραση των λαών, λέω, ε, μπορεί να ε, υποκύπτει σε πολυεθνικές σε ανάγκες, σε πολυεθνικά, αλλά όχι παγκόσμια και καθολικά συμφέροντα και να οδηγεί σε μια ομοιόμορφη οικονομική εξουσία που υπηρετεί άγνωστες εξουσίες. Αυτή είναι μια πρόκληση που πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική το να δώσουμε ε, ελπίδα στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι θα αναγνωρίσουμε την ανθρωποκεντρικότητα. Σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ικανότητες των ανθρώπων. Επομένως, ακριβώς σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επενδύσουμε. Ε, σε αυτά τα νέα ταλέντα τα οποία θα πρέπει να αναπτυχθούν και να καρποφορήσουν. Και βεβαίως το πρώτο σκέλος ε, είναι αυτό της εκπαίδευσης. Ξεκινώντας από την οικογένεια που είναι ε, το ουσιώδες κύτταρο και το οποίο δεν είναι δυνατό δυνατόν να διχοτομηθεί. μια ενωμένη οικογένεια η οποία έχει όλα τα θεμελιώδη στοιχεία που μπορούν να δώσουν ελπίδα στο μέλλον. Χωρίς μια τέτοια αλληλεγγύη τελικά ε, κατασκευάζουμε οικοδομήματα στην άμμο με τεράστιες κοινωνικές ε, ε, με τεράστιες ε, κοινωνικές επιπτώσεις. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η σημασία της ε, οικογένειας βοηθάει όχι μόνο τις επόμενες γενιές ε, αλλά και τις παλαιότερες, τους πολλούς ηλικιωμένους που συχνά ζουν χωρίς την οικογενειακή θαλπορή, χωρίς τη θαλπορή της οικογενειακής εστίας που τους συνοδεύει ή τους στηρίζει. Εκτός από την οικογένεια βεβαίως υπάρχουν και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα σχολεία και τα πανεπιστήμια η εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί στην παροχή τεχνικών γνώσεων αλλά θα πρέπει να ευνοήσει ε, μια, ε, ε, μια πιο περίπλοκη διαδικασία ανάπτυξης του ανθρώπινου όντως στο σύνολό του. Οι νέοι σήμερα απαιτούν μια πιο προσαρμοσμένη προς το μέλλον εκπαίδευση Πολλές επίσης ε, είναι και οι δημιουργικές ικανότητες ε, της Ευρώπης ε, σε πολλά θέματα της επιστημονικής έρευνας. Και βεβαίως αρκεί κανείς να σκεφτεί τις εναλλακτικέ μορφές ενέργειας που πραγματικά μπορούν να οδηγήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Η Ευρώπη πάντα ε, βρισκόταν στην πρώτη γραμμή ε, σε μια αξιοθαύμαστη δέσμευση όσον αφορά την οικολογία. Αυτή η γη μας πραγματικά χρειάζεται διαρκείς φροντίδες και διαρκή προσοχή και ο καθένας μας έχει προσωπική ευθύνη ε, να ε, ε, προστατέψει το δημιούργημα το οποίο βρίσκεται στα χέρια των ανθρώπων. Αυτό αφενός σημαίνει ότι η φύση είναι βεβαίως στη διάθεσή μας, μπορούμε να την απολαύσουμε και να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Από την άλλη όμως σημαίνει ότι δεν είμαστε τα αφεντικά της και οι κυρίαρχοι. Την προστατεύουμε, δεν είμαστε οι κυρίαρχή της. Επομένως ε, θα πρέπει να την ε, σεβόμαστε. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε αυτήν την αλαζονία ε, της ε, εξουσίας και θεωρούμε ότι μπορούμε να την χειριστούμε όπως θέλουμε. Δεν την προστατεύουμε, ε, δεν την χρησιμοποιούμε σωστά, τη χρησιμοποιούμε σαν να είναι η ιδιοκτησία μας, την οποία δεν χρειάζεται να θεραπεύσουμε και δεν χρειάζεται να προσέξουμε. Θα πρέπει όμως να τη χρησιμοποιήσουμε για το καλό και την έχουμε χρησιμοποιήσει και για το καλό. Αναφέρομαι εδώ στην ε, Γεωργία, ε, η οποία καλείται να θρέψει εκατομμύρια ανθρώπους που αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο πεθαίνουν από την πείνα, ενώ ε, τόνοι, εκατομμύρια τόνοι πετιούνται τροφίσε, πετιούνται κάθε μέρα από το καθημερινό μας τραπέζι. Πρέπει να σεβαστούμε ε, την φύση, ε, μην λησμονώντας ότι ο ίδιος ο άνθρωπος ε, είναι το κέντρο αυτής της γης και πέρα από την περιβαλλοντική οικολογία υπάρχει και η οικολογία η κοινωνική. Το δεύτερο πλαίσιο στο οποίο τα ανθρώπινα ταλέντα αναπτύσσονται είναι η εργασία. Θα πρέπει πλέον να βρεθούν και να ευνοηθούν οι πολιτικές απασχόλησης, αλλά κυρίως θα πρέπει να δοθεί ξανά αξιοπρέπεια στην εργασία, έτσι ώστε ε, να ε, προχωρήσει και να εξελιχθεί σωστά. Αυτό σημαίνει, από τη μία πλευρά, ότι θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι για να συνδυαστεί η ευελιξία της αγοράς ε, με την ανάγκη σταθερότητας και ασφάλειας όσον αφορά τις εργασιακές προοπτικές οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανθρώπινη ανάπτυξη των εργαζομένων. Απ' την άλλη πλευρά σημαίνει ότι θα πρέπει να ευνοηθεί ένα κατάλληλο κοινωνικό πλαίσιο το οποίο στόχο δεν θα έχει την εκμετάλλευση των ανθρώπων αλλά στόχο θα έχει να εγγυηθεί μέσω της ε, εργασίας η δυνατότητα να οικοδομηθεί η οικογένεια και να εκπαιδευτούν τα παιδιά. Ομοίως είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί το θέμα της μετανάστευσης. Δεν είναι δυνατόν να ανεχθούμε η Μεσόγειος να είναι ένα μεγάλο νεκροταφείο. Sui balconi che giungo σε αυτές ε, τις ε, βάρκες οι οποίες καθημερινά ε, φτάνουν στις ακτές της Ευρώπης υπάρχουν άνδρες και γυναίκες, άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται υποδοχή και βοήθεια η έλλειψη ε, μιας αμοιβαίας υποστήριξης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κινδυνεύει να ε, οδηγήσει σε λύσεις οι οποίες θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα ακριβώς γιατί είναι μεμονωμένες και δεν λαμβάνουν υπόψη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των μεταναστών η Ευρώπη θα πρέπει να έχει πλέον την ικανότητα, την δυνατότητα να αντιμετωπίσει όλες τις ε, προβληματικές ε, οι οποίες ε, συνδέονται με την μετανάστευση. Θα πρέπει με σαφήνεια να μπορέσει να προωθήσει την δική της πολιτική, συγγνώμη, πνευματική ταυτότητα και θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να τολμήσει να πάρει τις κατάλληλες νομοθετικές διατάξεις οι οποίες ε, θα δώσουν την δυνατότητα καλύτερα να υποδέχεται τους ε, μετανάστες. Ε, θα πρέπει να, δώσει αυτές, να αναλάβει αυτές τις σωστές πολιτικές οι οποίες θα είναι και θαραλέες έτσι ώστε να δώσει την δυνατότητα να βοηθηθούν οι μετανάστες στις δικές τους χώρες. Θα πρέπει να δράσουμε στα αίτια και όχι στα αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ε, συνείδηση της ταυτότητας είναι απαραίτητη έτσι ώστε να ε, ξεκινήσει κανείς διάλογο ε, και με συγκεκριμένες προτάσεις προς τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει στο μέλλον ε, να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι σε χώρες της Βαλκανικής, των οποίων η είσοδος στην Ευρώπη θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο ιδεώδες της ειρήνης μιας περιοχής η οποία πολύ έχει υποφέρει από σειράξει στο παρελθόν. Τέλος, ε, η συνείδηση της ε, δικής μας ταυτότητας είναι απαραίτητη στις σχέσεις με ε, τις άλλες γειτονικές χώρες, κυρίως αυτές οι οποίες βλέπουν την Μεσόγειο και οι οποίες πιέζονται από τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό και από την διεθνή τρομοκρατία εσείς ε, ως νομοθέτες θα πρέπει να αναπτύξετε και να διατηρήσετε την ευρωπαϊκή ταυτότητα έτσι ώστε οι πολίτες να ξαναβρούν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς της Ευρώπης αλλά και στη διαδικασία ειρήνης και ε, ε, ε, φιλίας που αποτελεί τη βάση του γνωρίζοντας ότι όσο πιο αναπτύσσεται η δυνατότητα των ανθρώπων τόσο περισσότερο διευρύνεται και η ατομική αλλά και συλλογική τους ευθύνη. Σας παρακαλώ λοιπόν κάνω έκκληση να εργαστείτε έτσι ώστε η Ευρώπη να ξαναβρει την καλή της ψυχή ανώνυμος συγγραφέας του δεύτερου αιώνα έγραψε ότι οι χριστιανοί αντιπροσωπεύουν στον κόσμο αυτό που η ψυχή αντιπροσωπεύει για το σώμα. Εσείς θα πρέπει λοιπόν να φροντίσετε και το σώμα και την ψυχή. Θα πρέπει να διατηρήσετε ε, την ιστορική μνήμη που είναι μια ε, ε, ιστορία πολλών χιλιετιών που αφορά και την Ευρώπη και τον χριστιανισμό. Πρόκειται για μια ιστορία στην οποία και λάθη υπήρξαν και αδικίες και σειράξεις αλλά παρόλα αυτά έδειξε πάντα επιθυμία να οικοδομήσει με βάση περάσει το καλό. Το βλέπουμε στην ε, ομορφιά των ε, χωρών μας, στην ομορφιά των πόλεών μας, το βλέπουμε ε, και στις διάφορες, στα διάφορα φιλανθρωπικά έργα τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε ολόκληρη την Ήπειρο. Αυτή είναι η Ευρώπη μας, αυτή είναι η ταυτότητά μας και η Ευρώπη χρειάζεται να ξαναβρει αυτό το ξεχασμένο της πρόσωπο έτσι ώστε να αναπτυχθεί σύμφωνα με το πνεύμα των πατέρων ιδρυτών, ειρήνη και ομόνια. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, έφτασε η ώρα να οικοδομήσουμε μαζί την Ευρώπη η οποία δεν θα στρέφεται γύρω από την οικονομία, αλλά θα στρέφεται γύρω από την αγιότητα του ανθρωπίνου όντως ε, και από τις ε, αναπαλωτρίωτες αξίες. να χτίσουμε μαζί την Ευρώπη η οποία ε, εναγκαλίζεται με θάρρος το παρελθόν της και κοιτάει με εμπιστοσύνη το μέλλον της, ε, ζώντας όμως πλήρως και με ελπίδα το παρόν της. Έφτασε η στιγμή να εγκαταλείψουμε την ιδέα μιας φοβισμένης Ευρώπης που αμφαλοσκοπεί και να ε, οδηγηθούμε σε μια Ευρώπη που θα πρωταγωνιστεί στην τέχνη, στην μουσική, στις ανθρώπινες αξίες αλλά και στην πίστη. Μια Ευρώπη η οποία θα στρέφεται προς τον ουρανό ε, και θα ακολουθεί τα ιδεώδη της. Ευρώπη, μια Ευρώπη η οποία θα περπατάει στη γη ε, με σταθερότητα και ασφάλεια και θα αποτελεί ε, μια πραγματικά, ένα πραγματικά πολύτιμο σημείο αναφοράς για όλη την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι κυρίε και κύριοι, το χειροκρότημά σα έδειξε ότι ο Πάπας Φραγκίσκος ε, σα άγγιξε. Είχα την εντύπωση ότι άγγιξε τις καρδιές όλων. Είμαστε ευγνώμονε και για την ομιλία σας αυτή, αλλά και για την τόσο μεγάλη ενθάρρυνση αυτό που είπατε εγώ το ε, εκλαμβάνω ως ενθάρρυνση να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο δρόμο που χάραξε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είναι ένας δρόμος που οδηγεί σε ένα καλό μέλλον. Μας δώσατε σημαντικές ε, συμβουλές και σας ευχαριστώ εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Είστε μια προσωπικότητα που δίνει προσανατολισμό ε, σε καιρούς που έχει χαθεί ο προσανατολισμός. Γι' αυτό σας είμαστε απείρως ευγνώμονες πρώτον που ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας απευθύνατε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι που ε, υποστηρίξατε τον Άγιο Πατέρα με την παρουσία σας και με ε, το χειροκρότημά σας, τον επιδοκιμάσατε. Νομίζω ότι έχουμε πολλά κοινά καθήκοντα και θα μας βοηθήσουν τα λόγια του Παπά Φραγκίσκου. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε στο Κοινοβούλιο.